liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten... Αγαπητοί κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω πως θα πρέπει να ξεκινήσουμε στην ώρα μας. Οπότε πρωτού περάσουμε στην ημερήσια διαταξή. Η συνάδελφος Κώστα ζήτησε το λόγο, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μόνο να πω σύντομα. Σήμερα πέρασαν δύο χρόνια από το τραγικό θάνατο των τριών φοιτητριών ε, του Εράσμου στην ε, Ισπανία, 13 λαμπρά παιδιά, κορίτσια που έχασαν τη ζωή τους, όταν έκαναν ε, με εκδρομή στην Βαλένσια. Ελίζα, Μοκίνα, Κλόε, Βερόνικα, Τζούλια, Κριστίνα, Πουόν Αν. Ήταν τα ονόματα των κοριτσιών. Εφτά ήταν Ιταλίδες, Γερμανίδα, Ρουμάνα, Αυστριακή, Γαλλίδα, και μία από το Σμπεκιστάν. Να πω ότι είναι παρόντες εδώ και κάποιοι φίλοι των συγγενών των θυμάτων. Είμαστε σε στενή επαφή με τις οικογένειες, εγώ από καιρό. Είμαστε κοντά τους, δείχνουμε αλληλεγγύη και ευχόμεθα το ταχύτο δυνατό να ολοκληρωθεί μια διαδικασία που κράτησε δύο χρόνια. Αλλά ακόμα δεν έχει δώσει πλήρη ικανοποίηση όσον αφορά τις οικογένειες, δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Με συγχωρείτε, λίγο ησυχία. Να επιθυμίσω κάτι. Ότι στην Επιτροπή Αναφορών υπήρξε αναφορά ενός νέου φοιτητή που ζήτησε κάτι σωστότατο. Να εναρμονιστούν στην Ευρώπη οι κανόνες για τις ασφάλειες, κυρίως όταν χάνεται μια ζωή και υπάρχει τόση μεγάλη επικοινομορφία, αυτό που καταβάλλεται να αποσυμίσει τι οικογένειε των σκανδαλώδε. και θα πρέπει να ληφθεί υποχρέωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κλείνω. Επρόκειτο περί μια εκδρομή που συνδεόταν όμω με το έρασμο, την εμπειρία έρασμο και θα πρέπει να παγκρυπνούμε για το επόμενο πρόγραμμα και στη διαχείριση του προγράμματο να υπάρχουν τα αμέγιστα εχέγγυα και η ασφάλεια όσον αφορά τα μεταφορικά μέσα που συνδέονται με τι δραστηριότητε ε, του έρασμο, που συνδέονται με το έρασμο. Μία σκέψη λοιπόν για εκείνου και για τι οικογένειέ του. Ε, γι' αυτό ήθελα να μιλήσω. Σε ευχαριστώ θερμά, Σίλβια που μας επενθύμησε σε αυτό το τραγικό δυστύχημα για ότι μας αποσαφήνισες ποια είναι τα διδάγματα που θα πρέπει να αντλήσουμε από αυτό για το μέλλον. Περνάμε τώρα στις ε, ψηφοφορίες. Ε, έχουμε ε, ε, μία πρόταση ψηφίσματος και μία γνωμοδότηση επί των οποίων θα ψηφίσουμε σήμερα. Ξεκινούμε λοιπόν με τη γνωμοδότηση ό,τι αφορά την έκθεση πρωτοβουλία, σε ό,τι αφορά την 7η έκθεση Τη επιτροπή σε ό,τι αφορά την ενίσχυση τη οικονομική κοινωνική και εδαφική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Διάκονο ήταν ο εισηγητής μα σε σχέση με αυτό το σημείο. Δεν ξέρω αν θέλει να πάρει το λόγο πρωτού ξεκινήσουμε με την πληροφορία. Όχι, τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε απευθεία. Ξεκινώ λοιπόν με την τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. Στο συγγνώμη. 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1, σε ό,τι αφορά την 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Σομβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 31. Το δεύτερο τμήμα της 31. Υπέρ, κατά, αποχές θα ήθελα να την ελέγξουμε. Την τροπολογία 31 λοιπόν, το δεύτερο τμήμα της, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται λοιπόν. 15 ψήφους υπέρ και 9 κατά. Έγινε μια παρέμβαση εκτό μικροφώνου. Ο πρόεδρο ε, λέει ότι ακόμα και αν είχε ψηφίσει δεν θα αλλάζει τίποτα στο αποτέλεσμα. Περνάμε στη 18 υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχέ. Θα ήθελα να ελέγξουμε και πάλι την 19 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. 19? Είμαστε 19 πάντα. Good. Jetzt geht's. Good. Ωραία, λειτουργήσε τώρα το μηχάνημα. Απορρίπτεται λοιπόν με 15 ψήφους κατά. 20 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές θα ήθελα να το ελέγξουμε, το δεύτερο τμήμα. Νομίζω πως απορρίπτεται, αλλά θέλω να σιγουρευτώ. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέραση τη ψηφοφορίας. 15 ψήφοι κατά, 11 υπέρ, απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω πως και αυτή απορρίπτεται, αλλά και αυτή θα ήθελα να την ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέραση τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται με 16 ψήφου κατά. 33 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Και την 33 να την ελέγξουμε. Νομίζω πω και αυτή απορρίπτεται. πάντα καλύτερα να σιγουρευόμαστε. Μάλλον η ίδια πλειοψηφία θα απορρίψει. 16 υποψήφοι λοιπόν κατά, 11 υπέρ, πράγματι απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προφορική τροπολογία 2 σε ό,τι αφορά την τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην ψηφοφορία επί του συνόλου της νομοδότησης. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται λοιπόν ηλεκτρονικά. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ, καμία ψήφο κατά και τέσσερις αποχές. Τα θερμά μας λοιπόν συγχαρητήρα στον εισηγητή. Και ελπίζουμε βέβαια πως η, επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή θα λάβει υπόψη τη δική μας γνωμοδότηση. Περνάμε τώρα στην πρόταση ψηφίσματος σε συνέχεια μια προφορική ερώτηση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια, πορεία των εργασιών και παρακολούθηση. Και εδώ ε, βασιζόμαστε βέβαια ε, στην διάσκεψη σε ό,τι αφορά την διαδικασία της ε, Μπολόνια των συμμετεχουσών χωρών τον Μάιο στο Παρίσι και θα ήθελα σε αυτό το πλαίσιο να στήσω από όλους τους συντονιστές να απευθυνθούν στους επικεφαλείς των πολιτικών τους ομάδων γιατί η ΣΥΟΠΗ δεν έλαβε καμία απόφαση τον τελευταίο καιρό σε σχέση με οποιαδήποτε προφορική ερώτηση, ε, με αποτέλεσμα να έχει υπάρξει μια συσσόρευση τώρα αιτηματών. Οπότε ε, παρακαλώ να εξηγήσετε στους επικεφαλείς ότι θα πρέπει οπωσδήποτε μέσα στον Απρίλιο να εγκριθεί αυτό το ψήφισμα, γιατί το Μάιο θα λάβει η χώρα διάσκεψη. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα έχει νόημα καν να εγκρίνουμε αυτό το ψήφισμα. Οπότε σας παρακαλώ να έρθετε σε επαφή με τους επικεφαλείς των πολιτικών σας ομάδων για να εξηγήσετε τη σημασία του να περάσει αυτό το ψήφισμα στην επόμενη Ολομέλεια. Θα ήταν κρίμα δηλαδή, γιατί θα χαθούν ε, όλες αυτές τις εργασίες που κάναμε στο πλαίσιο αυτού του ψηφίσματος. Νομίζω πως μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ξεκινούμε με τη συμβαστική τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 23. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 4 Ας ελέγξουμε, ας ελέγξουμε λέει πρώτος την 24. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την 24. Για την 24 λέει πρώτος, όχι τη συμβαστική τροπολογία 4. Ελέγχουμε την τροπολογία 24. Πέραση ψηφοφορία. 14 ψήφοι κατά, λοιπόν 11 υπέρ. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 30 υπέρ, κατά, αποχές, ας ελέγξουμε την 30, ηλεκτρονικά. Πέραση της φοφορίας, απορρίπτεται με 14 ψήφους κατά και 12 υπέρ. Περνάμε στην τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω πω απορρίπτεται με την ίδια πλειοψηφία, αλλά στο το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ελέγχουμε λοιπόν την τροπολογία 31. Πέρας. Όχι, εγκρίνεται με 13 ψήφους υπέρ και 12 κατά. Καλά λοιπόν που το ελέγξαμε. 32 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως απορρίπτεται, αλλά στην ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία για τη 46. Πέρας. Απορρίπτεται λοιπόν με 13 ψήφους κατά και 13 υπέρ. Περνάμε στην τροπολογία 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 51 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά χες εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 και τροπολογία 5 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές θα ήθελα να την ελέγξουμε την τροπολογία 7 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά πέρας απορρίπτεται με 13 ψήφους κατά και 13 ψήφους υπέρ τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα γιατί δεν σηκώσατε ψηλά τα χέρια οπότε ελέγχουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 11 πέρας εγκρίνεται με 18 ψήφους υπέρ και 7 κατά. Γι' αυτό σας παρακαλώ να σηκώνετε ψηλά τα χέρια για να τα βλέπω. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 15, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 16, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 17, υπέρ, κατά αποχές. Θα ήθελα να την ελέγξουμε, την 17 λοιπόν ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται με 12 ψήφους υπέρ και 11 κατά. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές, να την ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 18 γιατί υπήρξαν πολλές αποχές. Πέρασε της ψηφοφορίας. 15 ψήφι υπέρ, 7 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία για το σύνολο της πρότασης ψηφίσματος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της Εγκρίνεται λοιπόν με 23 ψήφους υπέρ και μία ψήφο κατά. Σας ευχαριστούμε θερμά και ελπίζουμε πως μέσα στην επόμενη όλο ε, μέλειά μας θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτή την πρόταση. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος ε, των ψηφοφοριών και περνάμε στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης. Σας παρακαλώ όσοι επιθυμείτε να εγκαταλείψετε την αίθουσα να το κάνετε με ησυχία. Ήσυχα και γρήγορα να εγκαταλείψετε την αίθουσα. Έχουμε λοιπόν το σχέδιο έκθεση για την ισότητα των γλωσσών ε, στην ψηφιακή εποχή. Η συγγήτρια Παρακαλώ, λίγη ησυχία. Λοιπόν, εξέταση σχεδίου έκθεση για την ισότητα των γλωσσών στην ψηφιακή εποχή. Είναι εδώ η συγγήτρια η συνάδελφος Τζιλέβανς. Θα ήθελα να σας πω ήδη για την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών ότι είναι η 10η Απριλίου στις 2 το μεσημέρι. Έχετε δηλαδή χρόνο μέχρι τότε. Στις 16 Μαΐου θα ψηφίσουμε σε ό,τι αφορά αυτή την έκθεση ιδίας πρωτοβουλία. Κυρία Εύαν, έχετε την έκθεση, την, τον λόγο για να σας παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πολιτικούς μου συμβούλους και τους εμπειρογνώμονες. Με βοήθησαν πολύ και ευχαριστώ και τη γραμματεία για το έργο που επετέλεσε επί της μέχρι τώρα. Προσβλέπω συνεργασία με τους κοιόδης ηγητές. Κατά τις επόμενες φάσεις, δυστυχώς, χρειαστήκαν περίπου 7 μήνες για να ληφθεί μια απόφαση για την κατανομή των ευθυνών μεταξύ της Ήτρα και της ΚΑΛΤ σχετικά με την έκθεση. Μόλις δύο εβδομάδες είχα στη διαθεσή μου για τη σύνταξη εκθέσεως και μία από αυτές ήταν πράσινη. Δεν μπορούσα να συζητήσω από κοντά με τους κοιόδησος όπως τα ήθελα για να βοηθήσουν στη σύνταξη της εκθέσεως, όμως προσβλέπω σε στενή συνεργασία μαζί τους από τούδε και στο εξή. Ποια είναι η ιδέα της εκθέσεως. Προήλθε από έξοχη μελέτη. Δημοσιεύτηκε από τη ΣΤΟΑ τον Μάρτιο πέρσι. Εκεί τονίστηκαν τα διάφορα προβλήματα που δημιουργούνται από τους ρωσικούς φραγμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εργασιακή κινητικότητα, διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, εμπόριο, δημόσιες υπηρεσίες. Η μελέτη δείχνει ότι νέα, οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν προβλήματα μεν για εκείνους που χρησιμοποιούν πιο σπάνιες γλώσσες. Παρ' όλα αυτά, εκείνοι θα ωφελούνται περισσότερο από τις τεχνικές εξέλιξεις. Οπότε η τεχνολογία των γλωσσών μπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστούν οι γλωσσικοί φραγμοί. Εξετάζοντας την έκθεση, θα ήθελα να προωθήσουμε αυτή την ιδέα. Προσωπικά, από την εμπειρία μου στην Ουαλία, μπορώ να πω ότι μιλάμε μια μειονοτική γλώσσα, τα ουαλικά, που παλεύει. Έχουμε λογοτεχνία, μουσική, παιδεία. Χρησιμοποιείται εκεί, αλλά στην ψηφιακή εποχή μειονοτικέ γλώσσες, όπως τα ουαλικά, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν με τις μεγαλύτερες γλώσσες στο διαδίκτυο και κυρίως με τα αγγλικά ο κόσμος περνάει τόση ώρα σχεδόν σε αγγλόφωνο ψηφιακό κόσμο και νέες τεχνολογίες όπως η Siri και η Alexa αλλάζουν τον κόσμο τον οποίο ζούμε αλλά δεν υπάρχουν αυτά τα προγράμματα στις μειονοτικές γλώσσες. Δεν είναι μόνο πρόβλημα των μειονοτικών γλωσσών. Πολλές γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αυτό το πρόβλημα. Ε, δηλαδή, μία μεγάλη γλώσσα, πλειοψηφική γλώσσα στον πραγματικό κόσμο, πάνει μια ψηφική γλώσσα στον ψηφιακό κόσμο. Η μελέτη έδειξε ότι κάποιε ευρύτατα ομιλούμενε γλώσσε, όπω εστονικά, λατωνικά, λιθουανικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν το ίδιο επίπεδο στήριξη από την τεχνολογία ή σε κάποιε περιστάσει λιγότερη υποστήριξη από ό,τι μειωνοτικέ γλώσσε, όπω είναι τα ουαλικά και τα βασκικά. Τα αγγλικά είναι η ευρύτερα ομιλούμενη γλώσσα στο διαδίκτυο Κυρίως αυτός οφείλεται στην επιρροή των Αμερικανικών φορέων, αλλά μεγάλο ποσοστό ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσης, 100% δεν μιλάει αγγλικά, δεν χρησιμοποιεί αγγλικά και υπάρχουν διαφορές μεταξύ ε, χωρών. Ισπανία, Ουγγαρία, Ισπανία και Βουλγαρία λιγότερο από το 20% του πληθυσμού μιλάει τα αγγλικά. Άρα δεν αφορά το πρόβλημα μόνο μειονοτικές γλώσσες, επηρεάζει όλους μας. Η έκθεσή μου εξετάζει το πώς οι πολιτικές Ευρωπαϊκής Ενώσεως μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση αναπτύσσοντας γλωσσικές τεχνολογίες σε μικρότερες γλώσσες. Είναι κρίσιμο λοιπόν να θεωρήσουμε ότι η τεχνολογία δεν είναι κίνδυνος και απειλή, αλλά ε, ένα μέσο διευκόλυνσης αντιμετωπίσης του προβλήματος. Η έκθεση υποδιαιρείται σε πέντε τμήματα. Ε, καταρχάς, εξετάζω τα εμπόδια για την επίτευξη ε, της γλωσσικής ε, υποβοήθησης στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ γλωσσών. Μετά προτείνω τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την τεχνολογία των γλωσσών, να στηρίζεται η γλώσσα από την τεχνολογία, οπότε να υπάρχει και η πολυγλωσσία που θα μπαίνει στο χαρτοφυλάκιο επιτρόπου, και είναι σημαντικό αυτό, αν θέλουμε να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίνεται στα προβλήματα που δημιουργούνται από την πολυγλωσία. Τρίτο, υπάρχουν συστάσεις για ερευνητικέ πολιτικές, όπως το να γίνεται μακροπρόθεσμη, να υπάρχει χρηματοδότηση μακροπρόθεσμη για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία, η δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας γλωσσικής τεχνολογίας, όπου μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες, να συναθροίσουμε ανθρώπους και εμπειρογνώμονες του τομέα και ένα πρόγραμμα για ψηφιακή πολυγλωσία. Η έρευνα για τεχνολογία γλώσσας κυριαρχείται κυρίως από μη ευρωπαϊκούς ε, φορείς και πρέπει να αλλάξει αυτό, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να ηγηθεί όσον αφορά την έρευνα στον τομέα. Τέταρτον, η έκθεση κάνει συστάσεις για εκπαιδευτική πολιτική, να εξασφαλίσουμε ότι η επόμενη γενιά των Ευρωπαίων θα μπορεί να ηγείται στον τομέα των γλωσσικών τεχνολογιών, θα μπορούν να αναπτύξουν την κατανόησή τους και τη δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν από πολύ νωρί αυτές τις τεχνολογίες. Και τελικά υπάρχουν συστάσεις για ιδιωτικέ επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς σχετικά με το πώς μπορούν να χρησιμοποιούν τις γλωσσικές τεχνολογίες προς όφελός τους πώς οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να κερδίσουν από καλύτερες, καλύτερα εργαλεία όπως αυτόματη μετάφραση, ε, μετατροπή από κείμενο σε ομιλία, αναγνώριση ομιλίας, που διευκολύνει διασυνοριακό εμπόριο και βελτιώνει την κατάσταση που είναι κατακαιρματισμένη η ψηφιακή αγορά. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω, σε επίπεδο 100 μελών και σε χαμηλότερο επίπεδο, θα χρησιμοποιήσουμε υφιστάμενε τεχνολογίε για να μειώσουμε τι γλωσσικέ ανισότητε. Οπότε έχουμε περίπου 80 περίπου διαφορετικές γλώσσες στην Ευρώπη, ανισότητες γλωσσών. Αυτό είναι το πρόβλημα, το πραγματικό. Με σωστές πολιτικές μπορούμε να το λύσουμε, να χρησιμοποιήσουμε την πολυγλωσσία προς όφελος ε, όλων μας. Ευχαριστώ. Yeah, Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση της έκθεσης. Και τώρα περνάμε στους σκιώδεις εισηγητές τρία λεπτά το πολύ ο καθένα. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια γιατί πραγματικά μέσα στον περιορισμένο χρόνο που είχε στη διάθεσή της κατάφερε να καταρτήσει μια πάρα πολύ καλή έκθεση και περιμένω με ανυπομονησία να συνεργαστούμε για να τη βελτιώσουμε, γιατί επειδή έχετε βελτιώσει, βέβαια, θέλω να τονίσω ότι τα εμπόδια τα οποία αναφέρατε και τα οποία συζητούνται μεταξύ των τρόπων Ήτρε και Κάλτα, δεν είναι κάτι τυχαίο. Γίνεται λόγο ακριβώς επειδή το θέμα έχει να κάνει με έρευνα, τεχνολογία και πολιτισμό. Και είναι πάντοτε δύσκολο να κάνουν το διαχωρισμό. Είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και πρέπει να το μελετήσουμε σε βάθος. Δεν θα επισέλθω τώρα σε λεπτομέρειες, πολύ ε, διεξοδικά. Μας τα εξήγησε και η συγγήτρια και συμφωνώ με την, προσωπική, με την προφορική της παρουσίαση σήμερα το πρωί. Θέλω όμως να πω ότι η εκθέση αυτή δεν βγαίνει από το πουθενά. Είναι μια πρωτοβουλία από κάτω προς τα πάνω. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 2012 το MetaNet για τις τεχνολογίες των γλωσσών, αυτή η πλατφόρμα, έκανε μια έρευνα και μια ανάλυση σε ό,τι αφορά την κατάσταση των γλωσσικών αυτών τεχνολογιών. Υπάρχει πράγματι ένα χάσμα μεταξύ της αγγλικής και άλλων γλωσσών, μεγάλων χωρών, μικρότερες γλώσσες, μειονοτικές, λιγότερο χρησιμοποιούμενες. Αυτά ε, υπάρχει πραγματικά ένα μεγάλο χάσμα. Αυτά ήδη το 2012 έχουν περάσει πέντε χρόνια έκτοτε και βλέπουμε να διευρύνεται το χάσμα μεταξύ των αγγλικών και των υπόλοιπων γλωσσών. Και αυτό είναι το θέμα. με την εισηγήτρια είχαμε και εμείς ε, προτείνει να αναλυφθεί αυτή η πρωτοβουλία για τη διενέργεια της μελέτης. Αυτή λοιπόν η πρωτοβουλία κάτω από τα πάνω πρέπει να συνεχιστεί. Η μελέτη είναι ίσως η πρώτη φορά που μας δείχνει ε, πώς πρέπει να προχωρήσουμε με τη λήψη πολιτικών αποφάσεων στον τομέα αυτό. Χρειάζεται μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Οι Ισπανοί επιστήμονες προετοίμασαν αυτή την πάρα πολύ καλή μελέτη με την τελική ανάλυση όλων των θεμάτων και η έκθεση τώρα της κυρίας Εύανς αντικατοπτρίζει τα πορίσματα στα οποία κατέληξαν οι μελετητές. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε Εύχομαι κάθε επιτυχία στην εισηγήτρια και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα τοποθετηθεί δεόντως. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γιάννα Τούν. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστούμε την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε να εκφράσω κάποιε σκέψει. Στον τομέα τη γενική ψηφιοποίηση αναθεωρούμε την άποψή μα για τη χρήση των γλωσσών. Περίπου εδώ και 100-200 χρόνια η γλωσσική ποικιλομορφία είχε υποστεί μεγάλε δοκιμασίε. Οι εθνικέ κυβερνήσει ε, επέλεγαν να υποστήξουν μια-δύο επίσημε γλώσσε και μειωτικέ γλώσσε. Ε, κρυζώθηκαν, εξαφανίστηκαν ή πέθαναν φυσιολογικό θάνατο. Υπήρχε καλό λόγο για μια τέτοια πολιτική. Την αναλογική εποχή ε, δεν επιτρέπεται να παρέχονται όλες οι υπηρεσίες όλε τι γλώσσε. Ήταν οξύ το πρόβλημα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δύσκολο να γίνει σωστή επιλογή. Επίσημη γλώσσα επίση θεωρήθηκε σαν αναγκαίο κοινό εργαλείο επικοινωνία που χρειάζεται να δημιουργηθεί μια, ένα αίσθημα ενότητα του κράτου, του έθνου. Αν κάποιο δεν κατανοούσε τι διαταγέ στο στρατό ή κάποια δήλωση σε επίσημη γλώσσα, θεωρείται ένα πρόβλημα που δεν επέτρεπε την εκκρέση κοινών Λοιπόν, η ψηφιοποίηση υπηρεσιών επιτρέπει πολλές γλώσσες να μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς να είναι κάτι ταπανηρό και ένα αποτελεσματικό πρακτικό παράδειγμα. Στην πατρίδα μου, την Εστονία, που είναι γνωστή η πολιτική που χρησιμοποιείται, που είναι αυστηρή για τη γλώσσα. Προωθούμε όμως την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, να γίνονται δηλώσεις φορολογικές, ε, ηλεκτρονικά φερρυπίν, οι δηλώσεις μπορούν να συμπληρώνονται όχι μόνο στα εστονικά, αλλά αγγλικά ή ρωσικά, που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στη χώρα οι γλωσσες Ε, περιπλέκεται όμω η, η, η, δουλειά εκείνων που ασχολούνται με τα φορολογικά. Μέχρι τώρα χρησιμοποιήσαν όμω τα εστονικά. Ε, χρειάζεται νέα τεχνολογία να ρυθμιστούν τα προβλήματα. Τόνισε το πρόβλημα η συγγήτρια τη επέκταση τη ψηφιακή τεχνολογία. Σοβαρό θέμα αν η γλώσσα δεν χρησιμοποιείται στην ψηφιακή τεχνολογία, δεν έχει πιθανότητα να επιβιώσει στο μέλλον. Η Ευρώπη είναι τόσο υπερήφανη για τη γλωσσική πολυμορφία. Πρέπει να αντισταθμίσουμε, να αποζημιώσουμε τις μειονότητες ε, για τις αδικίες που έχουν υποστεί στα κράτη. Και η ψηφιοποίηση ε, μας δίνει μοναδική ευκαιρία για κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μία φράση ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές για τους στόχους. Δεν θα εξαλειφθεί το κενό μεταξύ αγγλικών και άλλων γλωσσών. Εγώ είμαι γλωσσολόγος, γνωρίζω, ασχολούμαι με τα γλωσσικά θέματα. Είναι κάτι που δεν είναι στους αγγλόφωνου. Είναι δολοφόνο γλώσσα τα αγγλικά και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε με άλλες γλώσσες τα αγγλικά, πολωνικά, εστονικά, λετωνικά. Δεν μπορεί, υπερτερεί η αγγλική γλώσσα. Δυστυχώς ε, φοβάμαι και εγώ ότι αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστώ τη Γιάννα Τούμ. Η Νιριάρα. Συμφωνώ με την προλαλή σα. Πολύ συχνά συζητήσαμε για τα αγγλικά που είναι η γλώσσα δολοφόνο. Και όμω εδώ όλοι μιλάμε αγγλικά, παρόλο που έχουμε μητρικέ γλώσσε. Και θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τη μητρική γλώσσα. Αν έχουμε δικαίωμα να τη χρησιμοποιούμε, τη χρησιμοποιούμε σε αυτή την επιτροπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω Τζίλα Εύαν και όλου αυτού που ενεπλάκησαν στη σύνταξη τη εκθέσεω για την ισότητα των γλωσσών στην ψυχιακή εποχή. Ο χρονισμό εκθέσεων σημαντικό, διότι η Επιτροπή γνωρίζει ότι σίγουρα αλλάζουν οι εποχές και τα πράγματα και το προφανέστερο παράδειγμα η αναλλαγή της ε, τεχνολογίας και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να στερνιστούμε είτε μας αρέσει είτε όχι. Αυτό είναι κάτι που θα παραμείνει. Η έκθεση επιδιώκει να καλύψει τη μεγαλύτερη ανισότητα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην Ευρώπη, που είναι η γλωσσική ανισότητα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κύριοι που χρησιμοποιούν περιφερειακέ γλώσσε, μειωνοτικέ γλώσσε, είναι κάτι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο για τον 21ο αιώνα. Υπάρχουν μειωνοτικέ γλώσσε που μιλούνται σε κάθε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ενώση, από Σάμι στα Σουηδικά, τα Ιρλανδικά, στην Ιρλανδία. Και ο σαν και εμένα είμαστε 55 εκατομμύρια, 10% του πληθυσμού τη Ευρώπη που χρησιμοποιούν αυτέ τι γλώσσε. Άρα πρέπει να περάσουμε τέτοια έκθεση. Ήρθε η ώρα οι τεχνολογικέ πρόοδοι είναι πρόσδεκτε, δεν πρέπει να απειλούν όμω τι λιγότερο χρησιμοποιούμενε σημειωτικέ γλώσσε. Η ψηφιακή εποχή μπορεί να είναι πλατφόρμα για να διαφυλάξουμε και να προωθήσουμε τι λιγότερο χρησιμοποιούμενε και περιφερειακέ σημειωτικέ γλώσσε. Λοιπόν, υποστηρίζω την έκκληση του σχεδίου εκθέσεως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, την πολυγλωσία θα αναθέσει σε κάποιον επίτροπο. Όμω πράγματι εγώ θα προχωρούσα και παραπέρα και θα έλεγα ότι θα πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητη υπηρεσία που θα συσταθεί από του θεσμού τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και η λειτουργία αυτή τη υπηρεσία θα είναι να δρά σαν διαμεσολαβητής πολιτισμικός και πολυγλωσσικός, ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίζει την πολιτιστική και πολυγλωσσική ισότητα και θα πρέπει να δημιουργηθεί μια τέτοια υπηρεσία, διότι αφορά πολλά οριζόντια θέματα. Άρα είναι απόλυτα λογικό κατά την άποψή μου να δημιουργηθεί μια τέτοια υπηρεσία. Κλείνοντας, θα ήθελα να, κάν, να αναφερθώ σε κάτι πολύ σημαντικό για το πώς χρησιμοποιούμε εδώ στο Κοινοβούλιο την ε, γλωσσική ε, ποικιλομορφία. Έχουμε 23 επίσημες γλώσσες Ευρωπαϊκής Ενώσης που χρησιμοποιούμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω τη δική μου γλώσσα, που είναι μία από τις 23 επίσημες γλώσσες. Και αυτό τι δείχνει, δείχνει ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να αναγνωρίσουμε και να σεβαστούμε την πολιτισμική και γλωσσική ποικιλομορφία μας. Προσλέπω σε περαιτέρω επαφές μαζί σου Τζιλ και με άλλους επί της προοδευτικής αυτής ε, εκθέσεως. Ευχαριστώ. Άλλοι ομιλητέ τώρα, πλήν οδόν. Δύο λεπτά θα έχει ο καθένας, παρακαλώ. Ζαμπίνα Φερχάιν. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Θέλω να υπογραμμίσω αυτό που είπαν ορισμένοι προλαλήσαντες. Φυσικά δεν μπορούμε να αλλάξουμε το να υπάρχει μια λίγκουα φράγκα στην οικονομία ή στην τεχνολογία και αυτή τη στιγμή αυτή η γλώσσα είναι η αγγλική ή τα μας αρέσει όχι, είναι ένα γεγονός. Και δεν θα μπορέσουμε να το αλλάξουμε αυτό όσα μέτρα και αν πάρουμε. Ε, μπορούμε εμείς να το αποφασίσουμε ποια θα είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται ως γλώσσα συνεδρίων ή ως επικοινωνιακή, επικοινωνιακό μέσο. Αυτή θα είναι τα αγγλικά γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Υπάρχει όμως τεχνολογία που μας δίνει δυνατότητες ό,τι αφορά στην Ευρώπη ε, το να επιβάλλουμε ή την αναγνωρίσουμε τις γλώσσες τις άλλες ως ισότιμες με την αγγλική. Η τεχνολογία είναι ε, πλέον μας δίνει μάλλον πολύ περισσότερες δυνατότητες από ότι κατά το παρελθόν. Και στο ό,τι το λεξιλόγιο ή άλλα μέτρα για να προωθήσουμε τις ε, μειονοτικές γλώσσες. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πού μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποια μέτρα και τι ε, τεχνολογικές ε, εξελίξεις μπορούν να προωθήσουν ε, τη γλωσσική πολυμορφία και την πολυγλωσσία. Και εκεί θα πρέπει να δώσουμε το βάρος. Ευχαριστώ. Η Σίλβια Κώστα. Ευχαριστώ πολύ τη συνάδελφο Τζιλ για τη σημαντική και ενδιαφέρουσα έκθεση και θα συμβάλλουμε όλοι να ε, τονίσουμε κάποιες πτυχές. Πιστεύω και εγώ ότι θα πρέπει να συμβιώσουμε με αυτή την ισορροπία μεταξύ μιας ε, διαδεδομένης γλώσσας όπως είναι αγγλικά, που το έχουμε φτωχύνει σαν γλώσσα για το θέμα του γλωσσικού πληρολισμού, είναι και το, αφορά και το θέμα του να φτωχύνουν οι γλώσσες. Η σωστή αξιοποίηση της πολυγλωσσίας είναι ένας από τους πυλώνες του πολιτισμικού ε, πλουραλισμού που πρέπει να επικρατήσει στην Ευρώπη και να γνωρίζει στην Ευρώπη. Αυτό το πετυχαίνουμε σύμφωνα στις προτάσεις που γίνονται. Να υπάρξει μια εμβάθυνση των μελετών και της εφαρμογή των γλωσσικών τεχνολογιών που έχουν περάσει εδώ και 30 χρόνια από τότε από τις προσπάθειες που γίνονται για αυτή τη τεχνολογία σε εθνές επίπεδο. Και μπορεί να, να επηρεάσει και την προσφορά, τον προγραμματισμό, που έχουμε στο διαδίκτυο. Μια εφαρμογή να χρησιμοποιούνται διάφοροι πόροι κοινοί σε διάφορες γλώσσες. Πρόσβαση και αναγνώριση φωνητική που να είναι σε πολλές γλώσσες. Μπορεί να εφαρμοστεί στρατηγική οριζόντια και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα βελτιωθεί έτσι η δυνατότητα και η ποιότητα της πολυγλωσσίας εφαρμοσμένης μέσω τεχνολογίας. Είναι σημαντικό και κάτι άλλο. Η κατάρτιση για τη γλωσσική τεχνολογία και στα μαθήματα των πανεπιστημίων, στα προγράμματα των πανεπιστημίων. Και συμφωνώ και με την πρόταση να υπάρχει ειδική ευθύνη όσον αφορά τις τεχνολογίες και την τεχνολογική πολυγλωσία και την τεχνολογία της γλώσσας στα πλαίσια Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό είναι σωστό, πρέπει να ανατεθεί σε έναν επίτροπο και θα πρέπει να γίνει και εκπαίδευση του προσωπικού σε οριζόντιο επίπεδο. Όπω έλεγε η Τζιλ Evans όμως, να καθορίσουμε και τους ελάχιστους γλωσσικούς πόρου. Με ενδιαφέρει πολύ. Μπορεί να εξηγήσει καλύτερα αυτή την έννοια ε, που θεωρώ ότι είναι χρησιμότατη. Σας ευχαριστώ. Έριξα ε, μόλις ε, τώρα μια ματιά και ο αρμόδιος επίτροπος κύριο Ναύρατσης είναι ο αρμόδιος πράγματι για την γλωσσική πλωμιμορφία. Υπάρχει λοιπόν επίτροπος που έχει αυτή την αρμοδιότητα. Κύριε Σοντροβά έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την συγχύτρια την κυρία Εύανς γιατί το κείμενο είναι πολύ σαφές. Αναφέρεται δηλαδή με σαφήνεια τόσο στους κινδύνους αλλά και στις ευκαιρίες ε, που δημιουργεί η σημερινή κατάσταση. Καθώς ε, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις γλωσσικές τεχνολογίες για την καλύτερη επικοινωνία αλλά και για παράδειγμα για τη βελτίωση της κατάστασης των ε, γλωσσών και για τη διδασκαλία τέτοιου είδους γλωσσών και υπάρχει ακριβώς και αυτή η πρόταση ε, για ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο σε ό,τι αφορά αυτές τις γλώσσες σε έναν επίτροπο όπως ε, ε, και τη δημιουργία μιας σχετικής πλατφόρμας. Μπορώ να συμφωνήσω με αυτές τις προτάσεις. δηλαδή, θεωρώ πως οι γλώσσες μας είναι εργαλεία επικοινωνίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόμαστε μια lingua franca, μια γλώσσα μέσω της οποίας θα επικοινωνούμε και νομίζω πως θα είναι τα αγγλικά, γιατί ήδη τη χρησιμοποιούμε, ήδη υπάρχει ορολογία, οπότε μπορώ να συμφωνήσω με κάτι τέτοιο. Ενώ από την άλλη, ωστόσο, πλευρά, η κάθε γλώσσα αντικατοπτρίζει τον ιδιαίτερο πολιτισμό ε, από τον οποίο προέρχεται. Οπότε θα πρέπει ενώ χρησιμοποιούμε τα αγγλικά να ενισχύουμε τις εθνικές γλώσσες γιατί αυτές οι γλώσσες εκπροσωπούν ακριβώς την, κουλτούρα του κάθε ε, λαού. Οπότε εάν θέλουμε να διατηρήσουμε την πολιτισμική μας ε, ε, πολυμορφία, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διατηρήσουμε και την γλωσσική μας ε, πολυμορφία. Αλλιώς τα πράγματα δεν θα παραμένουν τα ίδια. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, κύριε Ευχαριστώ. Υπόθηκε ότι ίσω η κοινή μα γλώσσα, η lingua franca, χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά. Γι' αυτό αποφάσισα να χρησιμοποιήσω τη μητρική μου, τα ουγγρικά. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την έκθεση Συμφωνώ απόλυτα με το περιεχόμενό της. Είναι σημαντικότατο να ασχοληθούμε με το θέμα. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Τιμπορ Ναύρασιτς πράγματι είναι υπεύθυνο για την πολυγλωσία και το γραφείο του έχει προσωπικό που εργάζεται από αυτού. Όμως υπάρχουν ελάχιστα προγράμματα πολυγλωσσικά που προωθούνται. Ελπίζω λοιπόν αυτή η έκθεση να αποτελέσει έναυσμα προσπαθίας να τονίσουμε περισσότερο την πολυγλωσία. Είναι σημαντικό οι γλώσσες μικρότερων χωρών να τύχουν μεγαλύτερης προσοχής στην ε, ψηφιακή εποχή και για τις μειονότητες αυτές οι γλώσσες, οι περιφερειακές γλώσσες πρέπει να τονιστούν περισσότερο στην παιδεία στις περιοχές τους διότι εκεί όπου μιλούνται οι ντόπιε γλώσσες είναι πολύ σημαντικό οι κοινότητε που είναι να κατανοούν τις γλώσσες. Εγώ που είμαι Ούγγλος δεν βλέπω να απαραίτητο να μιλήσω γαλλικά. Αλλά σε περιοχές που ζουν πολλές μειονότητες είναι καλό η κάθε μειονότητα να μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα της άλλης. Γι' αυτό Είμαι ικανοποιημένο για το ένα εκατομμύριο υπογραφές που συνελέγησαν για ένα πρόγραμμα πολυγλωσσίας, ούτω ώστε να μπορεί να θεσπιστεί μια νομοθεσία που στηρίζει τις μειονοτικές γλώσσες, να χρησιμοποιούνται αυτές στην παιδεία, στα ψηφιακά μέσα και αν δεν έχετε υπογράψει για το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να το κάνετε. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ, ε, κυρία Sí. Ε. Ευχαριστώ. Δεν είμαι πάρα πολύ λίγο ρομαντική για πολλά. Ούτε και με τις γλώσσες είμαι ρομαντική. Αντί να προστατεύσουν πρώτα απ' όλα τις μειονοτικές γλώσσες, καλύτερα να προστατεύσουν πρώτα τις μειονότητες που τις μιλάει. Και όχι να ενισχύουμε μόνο την κοινή γλώσσα τα αγγλικά. Ελπίζω να μην χαθείστε μετάφραση ε, μια φράση πολύ σημαντική που πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν ξέρω ποιος το είπε, κάποιος ε, ξακουστός φιλόσοφος. Η επιβολή μιας γλώσσας στις υπόλοιπες ε, δεν είναι ε, το χειρότερο. Το χειρότερο είναι να μην επιβληθεί καμία. Αυτό στο ένα σοφός. Έτσι λίγο για να... Είμαι ο δικηγόρος του διαβόλου, μάλλον, ο του διαβόλου. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μόργαν. Θα ήθελα να θέσω κάτι. Δεν θα επαναλάβω άλλα που υπόθηκαν. Χρειάζεται μια εγκάσια κοινή γλώσσα, είναι προφανές. Το θέμα που αναδύεται και θα αναδυθεί όταν θελοποιηθεί το Brexit είναι το εξή. Μήπως σαν επίσημη γλώσσα, να γίνει επίσημη γλώσσα η γλώσσα μιας χώρας που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι τέτοια κοινή γλώσσα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να τεθεί. Ναι, είναι ένα σαρπαστικό ερώτημα αυτό. Ο κύριο Μαλίνοφ έχει Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, η γλωσσική ισότητα ε, δεν θα πείτε αν μιλάμε όλοι αγγλικά. Εγώ θέλω να αναφέρω κάτι που δεν είναι ακριβώς ε, μέσα στην έκθεση. Ως εκπρόσωπος των κρατών, θέλω να πω το εξής. Εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει αναγνώριση των γλωσσικών ε, πιστοποιητικών και τίτλων γλωσσικών σπουδών. Υπάρχουν δυσκολίες και εμπόδια στην αναγνώριση αυτών των πτυχίων. Δεν υπάρχουν δομές σε κάποιες χώρες όταν αφορά αυτές ε, λιγότερο μιλούμενες γλώσσες. Τώρα το βλέπω αυτό το πρόβλημα Να έχουμε δηλαδή πολλούς που πηγαίνουν σε άλλες χώρες να κατοικήσουν και σίγουρα μαθαίνουν τη γλώσσα της χώρας, αλλά δεν υπάρχουν εγγύησει στο ότι θα μπορούσαν να μάθουν ή τέλο πάντων να έχουν κάποια και στη δική τους γλώσσα. Υπάρχει το British Council, υπάρχει το γέτε. χώρα υποδοχής που θα πρέπει να φροντίσει για την εκπαίδευση, τη γλωσσική. Νέες δυνατότητες προσφέρει νέα αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ. Äh, σα ευχαριστώ θερμά. Ε, να κάνω και εγώ μια παρατήρηση από τη δική μου πλευρά. Καταρχήν να σα ευχαριστήσω θερμά ε, για ένα πολύ ε, καλό κείμενο. Όπως καταδεικνύει η συζήτηση που έγινε πρόκειται για ένα πραγματικό πρόβλημα εδώ και θα ήθελα πραγματικά ε, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς δηλαδή, να λάβουμε υπόψη μας πιο σοβαρά αυτό το ζήτημα. Για παράδειγμα, πρόσφατα ε, χρειάστηκε πριν από λίγο καιρό να αποστείλω έτσι μια πολύ εμφατική επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέροντας ότι ακόμα και στο έκτο έτος του Erasmus Plus, οι σχετικές πληροφορίες στο νηστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμος μόνο στην αγγλική γλώσσα, τόσο σε ό,τι αφορά τις βασικές κατευθύνσεις δουλειών όσο και σε ό,τι αφορά τις περαιτέρω πληροφορίες. Σε ό,τι αφορά τις κατευθύνσεις μπορεί να βρει κανείς καμιά άλλη γλώσσα, για παράδειγμα τα γαλλικά, αλλά σε ό,τι αφορά ε, τις μικρότερες γλώσσες δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Ε, η Επιτροπή απάντησε άμεσα και είπε ότι έγιναν βελτιώσει και βέβαια μέσα σε επόμενε εβδομάδε εγώ θα ελέγξω αν, κατα... αν πράγματι προέβησε βελτιώσει. Πάντω πραγματικά θεωρώ πω η γλωσσική πολυμορφία προωθείται μόνο μέσω τη διαθεσιμότητα ε, ε, όλων των εγγράφων ε, από τη δική μας πλευρά. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταδείξουμε ότι πραγματικά παίρνουμε στα σοβαρά αυτή τη γλωσσική πολυμορφία και ότι δεν επιθυμούμε να εξαφανιστούν οι μικρότερες γλώσσες. Θα πρέπει όλοι δηλαδή οι πολίτες μας να έχουν ίση πρόσβαση στις πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί υποχρέωσή μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναφέρουμε τα κακό σε κείμενα και όπου αυτό χρειάζεται να αποστέλουμε μία επιστολή στο αρμόδιο θεσμικό όργανο όπου θα προεγκαλούμε για την κατάσταση αυτή. Πολύ συχνά ε, βλέπουμε ότι ε, πληροφορίες ε, μπορεί να είναι διαθέσιμε σε τρεις γλώσσες, σε μία, αλλά σε καμία περίπτωση σε 24 και αυτό είναι αρνητικό. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. Εύχομαι κάθε επιτυχία στους σκιώδεις εισηγητές, αλλά είμαι απολύτως βέβαιο ότι θα φτάσουμε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και ελπίζω βέβαια πως ε, τελικά αυτή η πρόταση θα οδηγήσει και σε ε, ένα σχετικό αποτέλεσμα, αυτό που επιθυμούμε. Δεν ξέρω αν ο εκπρόσωπος της Επιτροπής θέλει να πάρει το λόγο. Okay. Dann vielen herzlichen Dank. Καλώς. Θα ξαναδώσω λοιπόν το λόγο στην ε, Jill Evans για να σχολιάσει τα όσα μόλις τώρα υπόθηκαν στη συζήτηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όλα τα σχόλια νομίζω ότι αντικατοπτρίζουν το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει σε αυτό τον τομέα και τη σημασία του θέματος και είμαι αισιόδοξη. Πιστεύω ότι με την έκθεση αυτή μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Είναι σημαντικό για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι σε ό,τι αφορά την επικοινωνία δεν μπορεί κανείς να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τον πλησίον εάν δεν μιλούν στην κυριολεξία όμως την ίδια γλώσσα. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό για το μέλλον της Ευρώπης. Και χαίρομαι ιδιαίτερα με τα σχόλια και την ανταπόκριση των συναδέλφων και περιμένω την πρώτη συνάντηση των σκιωδών, σίγουρα βέβαια και τις συμβολές όλων των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Προθεσμή κατάσταση τροπολογιών 10 Απριλίου, 2 το μεσημέρι και ψηφοφορία 16 Μαΐου. Επόμενο σημείο της μεσιάς διάταξης, το 11, είναι εξέταση μιας γνωμοδότησης για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, συγητής ο κ. Τζαμπάσκι. Προθεσμία κατάσταση τροπολογιών 26 Μαρτίου, 12 το μεσημέρι. 25 Απριλίου ψηφίζουμε. Η αρμόδια επιτροπή είναι ΑΦΚΟ, καθήλυνα αρμόδια ψηφίς 24. Παρακαλώ, κύριε Τζαμπάσκη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών είναι ένα τμήμα της Συνθήκης Λισαβόνας. Είναι καινοτόμο μέσο που ενθαρρύνει την άμεση δημοκρατία σε διεθνές επίπεδο και εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η αρχή της εν λόγω είναι να παρέχει στους πολίτες των κρατών μελών τη δυνατότητα να έχουν πρωτοβουλία. Ο μηχανισμός είναι περιπλοκότατος και μέχρι τούδε εμπειρία καταδεικνύει ότι χρειάζεται ριζική μεταρρύθμιση. Ευτυχώς το 2017, χάρη στο έργο της δικής μας Επιτροπής, της Επιτροπής Πολιτισμού και της ΑΦΚΟ, είχαμε κάποια αποτελέσματα. Και ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει. Ελήφθησαν υπόψη οι εκθέσεις και διάφορες μελέτες. Επίσης έγιναν διαβουλεύσεις και με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Αναμφισβήτητα η αναθεωρημένη πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσε να επιλύσει κάποια προβλήματα που διαπιστώσαμε με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών, όπως χαμηλότερο όριο ηλικίας για τους πολίτες που μπορούν να συμμετάσχουν σε κάποιες από τις πρωτοβουλίες. Αυτό θα αποτελούσε ένα σαφές μήνυμα για τη νέα γενιά που δεν ενδιαφέρεται τόσο για την πολιτική διαδικασία. Να τους δείξουμε ότι υπάρχει τρόπος να συμπεριληφθούν στη διαδικασία οι νεότεροι. Όμως θα πρέπει να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου διότι υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς που δεν έχουν επιληθεί στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως η άρνηση μειώσεως της απέτηση για ελάχιστο αριθμό 100 μελών που πρέπει να καλύπτονται για συμμετοχή σε πρωτοβουλία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει η έλλειψη συγκεκριμένου εργαλείου μέσω του οποίου μια επιτυχής πρωτοβουλία θα μπορούσε να μετατραπεί σε πρόταση νομικού περιεχομένου από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό προβλέπει το άρθρο 11.4 ε, της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρόν στόχος, ο πραγματικός στόχος είναι να έχουμε μια νομική πρωτοβουλία που θα προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα γίνεται αποδεκτή, θα απορρίπτεται από το Συμβούλιο ή το Κοινοβούλιο. Μόνο τέσσερις πρωτοβουλίες πολιτών πέρασαν το πρώτο στάδιο και γι' αυτό Θεωρώ ατυχές ότι δεν υπάρχει σχετική πρόταση να καλύψει το πρόβλημα ε, στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Ευχαριστώ κύριε Τζαμπάσκη. Περνάμε στους κοιόδες ηγητές. Κύριος Μαλίνοφ, με δύο λεπτά παρακαλώ το πολύ. Ξεκινάτε εσείς, ναι. Νομίζω ότι όλοι καλωσορίσουμε την πρώτη αναθεώρηση. Εγώ δεν ελπίζω, απλά είμαι βέβαιος ότι θα υπάρχει και τρίτη και τέταρτη αναθεώρηση πρωτοβουλίας. Ας δούμε λοιπόν την αναθεώρηση αυτή ως πρώτη θετική κίνηση και ίσως να μην περιμένουμε ότι θα είναι και πια ε, τόσο ριζική αυτή η αναθεώρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι Ένωση Δημοκρατιών. Βασίζεται στην ε, αρχή της ε, αντιπροσωπευτικότητας και είναι ότι πιο κοντά, αν μπορώ να το χαρακτήσω έτσι, στην άμεση δημοκρατία και νομίζω ότι αυτές τις νέες αλλαγές πρέπει να τις υποστηρίξουμε γιατί πηγαίνουν προς σωστή κατεύθυνση. Μπορεί κάποιες φορές ε, να έχουμε άλλου, άλλες αρνητικές ε, αλλαγές, τις οποίες δεν θα επιμείνω όμως. Ό,τι αφορά την ηλικία για τη συμμετοχή στη διαδικασία που από 18 πηγαίνει στα 16. Αν αυτό το δούμε από πρακτικής πλευράς, και επειδή η νομοθεσία σε πολλέ χώρε δίνει τη δυνατότητα στου νέου να ψηφίζουν από την ηλικία των 18 για κάποιου δραστήριου νέου στην Ευρώπη, μπορούν ε, για τι ευρωπαϊκέ πρωτοβουλίε να έχουν κάποια πολιτική δράση. Όσο δεν θα μπορούν δηλαδή ακόμη να είναι πολιτικά δραστήριοι στη χώρα του. Ε, και αυτό θα το θυμούνται όλοι στη ζωή. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση το να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα. Φυσικά μπορούμε να ασκήσουμε κριτική στην πρόταση ότι δεν είναι αρκετά τολμηρή, δεν πηγαίνει αρκετά μακριά, δεν είναι αρκετά ε, Ό,τι δεν αφορά τα στοιχεία πρέπει να παρέχουν οι πολίτες, έχουμε μια μείωση των στοιχείων. Και κάτι άλλο πολύ θετικό είναι η συμμετοχή βασίζεται στην εθνικότητα και όχι ε, και στον τόπο διαμονή. Αυτό είναι μια σημαντική βελτίωση γιατί έτσι περισσότερο κόσμο μπορεί να συμμετάσχει. Θα είναι πιο εύκολη η διαδικασία, ίσως δεν θα είναι τόσο γρήγορη. Οι αλλαγέ θα θέλαμε να ήταν πιο τολμηρέ. Εντάξει, πάντω πηγαίνουμε προ σωστή κατεύθυνση και είναι μια καλή βάση για την τρίτη αναθεώρηση που θα έρθει αναπόφευκτα, πιστεύω. σω σε κάποια χρόνια από τώρα, βέβαια. Ευχαριστώ, θα μιλήσω στα πορτογαλικά. Πράγματι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την αναθεώρηση, καθώς ε, βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει μια προσπάθεια και από την πλευρά τη Επιτροπή να υπάρξει μια αλλαγή, μια βελτίωση. Αυτή η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ε, Πολιτών ε, πρόκειται να βελτιωθεί με αυτή τη νέα πρόταση. Υπάρχουν δηλαδή κάποιε βελτιώσει, υπάρχει μια πλούστευση τη σχετική διαδικασία αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει η πρόταση να εστιάσει περισσότερο στη μείωση των δαπανών αλλά και στη μείωση των ε, γλωσσικών φραγμών που μπορούν να υπάρχουν σε ό,τι αφορά αυτέ τι ε, πρωτοβουλίε και στου οποίου φραγμού μόλι τώρα αναφερθήκαμε. Πράγματι δηλαδή θα πρέπει να στεφθεί επιτυχία αυτό το εργαλείο ε, αυξημένη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. θεωρώ πω είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει περισσότερη τεχνική και νομική υποστήριξη των πολιτών στο πλαίσιο αυτή τη διαδικασία της προσχώρησε μια τέτοια πρωτοβουλία και στο πλαίσιο, για παράδειγμα, ε, των, ε, της συγκέντρωσης των δηλώσεων υποστήριξης θα πρέπει να προσαρμόσουμε τον αριθμό αυτών των υπογραφών έτσι ώστε ε, να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα θα πρέπει παρόλα αυτά να υπάρξει, να, να συνεχιστεί η ευελιξία α, των σχετικών προτάσεων ε, γιατί σε ό,τι αφορά την έγκρισή τους, γιατί ήδη στην πρώτη φάση της καταχώρησής τους μεγάλο τμήμα των ε, πρωτοβουλειών απορρίπτεται από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα, ο διασυνοριακό ε, διάλογο σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και η δυνατότητα συμμετοχή των πολιτών περιορίζεται με αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη μία πλευρά θα πρέπει να ενημερώνει τους διοργανωτές τέτοιων πρωτοβουλειών σε ό,τι αφορά την ποιότητα των ε, προτάσεων τους και να τους δίνει τις δυνατότητες να το κάνουν. Ίσως ε, σε αυτό το ε, πλαίσιο να έχουμε βέβαια αναθέσει υπερβολικά πολλές αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να το αυτό. Θα πρέπει να ε, ε, εστιάσουμε περισσότερο στην συμμετοχική δημοκρατία, δηλαδή στην δυνατότητα των πολιτών να συμμετέχουν άμεσα σε τέτοιου είδου πρωτοβουλίε και τα συνέπεια στο πολιτικό γίγνεσθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Μαρία Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κύριο Ταμπάσκη για την γνωμοδότηση αυτή. Στόχο μα είναι η πρωτοβουλία αυτή να είναι ένα αποτελεσματικό δημοκρατικό εργαλείο για του Ευρωπαίου πολίτε. Τέσσερι μόνο πρωτοβουλίε, όπω ξέρουμε, έφτασαν ε, το όριο του 1 εκατομμύριου υπογραφών. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη απλούστευση τη διαδικασία και καλύτερη, μεγαλύτερη πληροφόρηση των πολιτών, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτικών. Χαίρομαι Ακούω ότι η πρόταση της Κομισιόν ε, περιλαμβάνει πολλές από τις υποδείξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως είναι η μείωση του κατώτατου όρου για την κατάσταση πρωτοβουλία ή η δυνατότητα την ε, ημερομηνία έναρξη ε, τη διαδικασία υπογραφών να την ορίζουν οι οργανώσει ή να δημιουργείται μια, ένα νομικό πρόσωπο για την κατάθεση μια πρωτοβουλία πολιτών. Πολίτες πρέπει να χρησιμοποιούν περισσότερο αυτό το εργαλείο. Συγγνώμη, έχετε και το τηλέφωνο μου ταυτόχρονα. Με τον κύριο Νταμπάς και συμφωνώ και εγώ ότι πέντε ε, θα να ο κατώτατο αριθμό ε, των ε, κρατών μελών που θα εκπροσωπούνται και θα πρέπει να στηρίξουμε αυτέ τι τροπολογίε. Καλύτερη επικοινωνία, στρατηγική επίση είναι κάτι απαραίτητο. Στην πρωτοβουλία αυτή να είναι πραγματικά αποτελεσματική και να προωθήσει ενεργού πολίτε που θα συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά δρόμενα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι σαφέ ότι θα πρέπει να κάνει περισσότερα πράγματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να εισακούει τι ανησυχίε των πολιτών. Βλέποντα αυτά που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δώσει κάποια συνέχεια στι πρωτοβουλίε πολιτών, διαπιστώνουμε ότι δεν έχουν γίνει και πολλά πράγματα. Μόνο τέσσερις πρωτοβουλίες πέρασαν τη διαδικασία και μόνο δύο ε, βρήκαν συνέχεια. Ξέρετε τι προσωπεύει αυτό. Να συλλέξει κανείς εκατομμύρια υπογραφές και μετά να μην δοθεί καμία συνέχεια στην πρωτοβουλία. Μπείτε στη θέση εκείνων που θέλησαν να συμμετάσχουν στη δημοκρατική αυτή διαδικασία και είδα να μην δίνεται καμία συνέχεια. Είναι αλήθεια ότι η πρωτοβουλία των πολιτών είναι ένα πολύ σημαντικό δημοκρατικό εργαλείο, αλλά βλέπω ότι ο απολογισμός είναι καταστροφικός. Φοβούμε ότι η αλλαγή η τροποποίηση των κανόνων θα καταστήσει δυσχερέστερη τη διαδικασία. Και θα δώσουμε μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν δεν θέλει να δώσει συνέχεια σε κάποια πρωτοβουλία πολιτών. Αν κατάγεστε από μια μικρή χώρα με 5 εκατομμύρια πληθυσμό Φερρυπίν, όπως είναι στη χώρα μου, τότε τα πράγματα δεν είναι ίσα όπως σε μεγαλύτερες χώρες. Θα πρέπει να ληφθεί ως υπόψη και αυτή η συνισταμένη. όταν γίνεται ένα διασυνοριακό διάβημα. Το βασικό είναι ότι αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών δεν έχει νόμιο παρά μόνο αν έχει κάποια αποτελέσματα, αν δοθεί κάποια συνέχεια σε μια πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. It's Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την, ε, τον εισηγητή ε, και απηχώ και εγώ τα σχόλια που ακούστηκαν. Υπήρξαν πολλές ελπίδες για την πρωτοβουλία των πολιτών όταν θεσπίστηκε αρκετά και κάποιες οργανώσεις ΜΚΟ και ομάδες ήταν ενθουσιώδεις στην αρχή. Απλούστευση λοιπόν είναι κρισίμου σημασίας, κυρίως η συμμετοχή των νέων είναι πάρα πολύ σημαντική. Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε να θαρρύνουμε τους νέους να συμμετάσχουν περισσότερο θα ήταν κάτι ευπρόσδεκτο διότι προσφέραμε αυτό σαν έναν τρόπο να συμμετάσχει ο πολίτης στις εργασίες, τη εργασίες Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε αυτό να το πετύχουμε με αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστώ. Κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μας καλέσατε και μας δίνετε το λόγο. Λουκ Μπότιγκαρτ, Είμαι αρμόδιος της μονάδας που ασχολείται με το θέμα. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες και τα σχέδια τροπολογιών. Τα εξετάσαμε και αυτά, τα στοιχεία. Κατανοώ ότι κάποια μέλη είπαν ότι κάποιες βελτιώσεις προτάθηκαν. Θέλω ακροθυγώς να τονίσω, κυρία Πρόεδρε, ποιος ήταν ο στόχος της αναθεωρήσεως. Βασικά στοιχεία της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποια ήταν να είναι πιο προσβάσιμη πρωτοβουλία των πολιτών, πιο εύκολο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους διαφόρους. Δεύτερος στόχος είναι να μπορεί να πετύχει τα πλήρη αποτελέσματα, εργαλεία για πρόθεση συζητήσεω και συμμετοχή πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η Ευρωπαϊκή Ένωση να πλησιάσει του πολίτε με αυτό το μέσο. Αυτή είναι η επίσημη στόχη. Απλούστερα να το θέσουμε. Η πρόθεση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το τονίζω, ότι η Επιτροπή Juncker έχει θέσει στόχο ότι ο μέγιστος αριθμός των πρωτοβουλειών που υποβάλλεται να μπορούν να καταχωρούνται καταρχάς και δεύτερον να έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να πετύχουν τη συλλογή τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου υπογραφών. Οι τελευταίες 17 πρωτοβουλίες που είχαμε στην Επιτροπή Juncker έπρεπε να απορρίψουμε μία που ήταν να σταματηθεί το Brexit. Και όλοι σε αυτή την αίθουσα θα δεχτούν ότι αυτό δεν ήταν στην εντολή και εξουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να το εφαρμόσει δυνάμει των συνθήκων και να επιτρέψει περαιτέρω δράση. Απέδειξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι πρόθυμη να κάνει επιτυχή την πρωτοβουλία των πολιτών, περισσότερο δε με την τρέχουσα πρόταση. Την ιτόριο ηλικία των 16 ετών, χαίρομαι που το τονίσατε αυτό. Οι πολίτες που δεν μπορούν ακόμα να εκφράσουν πολιτική άποψη σε εθνικό επίπεδο, αν κρατήσουμε το όριο των 16 ετών, θα μπορούν να κινηθούν πολιτικά και ο μέσος κύκλος πριν η αδίποτε πρωτοβουλία καρποφορήσει και τύχει περαιτέρω επεξεργασίας ε, είναι 18 μήνες. Όταν υποστήριξαν την πρωτοβουλία ήταν 16 κάποιοι και μέχρι να υπάρξει δράση οι άλλοι θα συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας. Άρα με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε 10 εκατομμύρια παραπάνω πολίτες που μπορούν να επηρεάσουν τα τεκτενόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά, προβλέπουμε μέτρα ενημέρωσης και βοηθείας. Θα κάνουμε και περισσότερα όμως, κυρίως μέσω της συλλογική αυτής πλατφόρμα που έχει προταθεί. Ευχαριστούμε το Ευρωκοινοβούλιο για τα πιλωτικά προγράμματα που μας δίνει την χρηματοδότηση κατέτοιου και 10 Απριλίου. Είναι οι μέρες της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, όποιος μπορεί να παρασταθεί. Ε, από την ΕΚΟΣΟΚ διοργανώνεται, την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή. Εκεί θα ξεκινήσει η πρώτη φάση της πλατφόρμας στο διαδίκτυο, να ενημερώσουμε τους πολίτες, να μπορούν να ανταλλάξουν οι πολίτες απόψεις, να συνεργαστούν πολίτες από 7 κάτι μέλη σε αυτή τη φάση για να διοργανώσουν κάποια εκστρατεία, να έχουν ιδέες περί χρηματοδοτήσεως, περί της ε, εγκαθίδης επικοινωνίας κλπ. Ελπίζουμε ότι αυτό θα προωθήσει περαιτέρω τις πρωτοβουλίες και να αυξηθεί ο αριθμό των πρωτοβουλειών που θα, φτάνουν, θα καταχωρούνται και θα συλλέγουν ένα εκατομμύριο υπογραφές. Κάτι που δεν αναφέρθηκε, αλλά συμπεριλαμβάνεται στις αλλαγές. Τι προτείνουμε. Μερική καταχώρηση να θεσπιστεί νομικός. Για την ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κάνει αυτό όταν δεν μπορεί να καταχωρηθεί πλήρης πρωτοβουλία θέλαμε τουλάχιστον μερικά να καταχωρούμε κάποια πρωτοβουλία. Είναι σημαντικό και τι προβλέπουμε. Και συμπαμβάνεται στην τροπολογία σας. Όταν αποστέλλετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για καταχώρηση πρωτοβουλία και αν θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν πρώτης, στην πρώτη ανάγνωση, ότι ίσως θα ήταν δύσκολο να καταχωρηθεί πλήρως, πάμε πίσω στους οργανωτές εντό μηνό, του ενημερώνουμε δεόντω. Αυτοί έχουν ένα μήνα να σκεφτούν κατά πόσο θέλουν να αναδιατυπώσουν την πρωτοβουλία του ή να αφαιρέσουν κάποια τμήματα αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαφώ δεν θα συγκράψει το κείμενο για αυτού. Δεν θέλουμε να παίξουμε το ρόλο, αλλά θα του δώσουμε συμβουλέ στο βαθμό που επιτρέπεται για το πώ μπορεί να βελτιωθεί η πρωτοβουλία και μπορεί να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα καταχώρηση. Το προβλέπουμε ήδη και σε κάποιε τροπολογίε λέτε ότι μετά θα μπορούν ακόμα να καταχωρήσουν εν μέρη το υπόλοιπο. Αυτό θα δημιουργήσει μεγαλύτερη ασάφεια, πιστεύουμε, και θα, αυξήσει τον αριθμό διοικητικών βημάτων. Δεν θα προσθέσει διαδικασία. Άρα, τι λέμε, μα στέλνουν την πρωτοβουλία, αν υπάρχουν ανησυχίε, τι τονίζουμε, το σκέφτονται, μα ένα μήνα μα το ξαναστέλνουν. Σε τρει μήνε, λοιπόν, θα επικρατήσει αφήνεια μέσω τη καταχωρήσεω. Βεβαίω, αν τα αρνηθούμε εξ ολοκλήρου ή εν μέρη, μπορούμε να στο δικαστήριο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπω είδαμε και σε πρώτερε υποθέσει. Θέλω να πω ότι είχαμε έξι υποθέσει που εξετάστηκαν από το δικαστήριο. Σε δύο υποθέσει το δικαστήριο είχε άλλη άποψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήταν κατά. Τέσσερι, 66% επιβεβαίωσαν τη θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι δηλαδή ότι προσπαθούμε να χειραγωγήσουμε το παιχνίδι, αντιθέτω. Προσπαθούμε να κινηθούμε σωστά. Δόξα τω Θεώ, στι 4 από 6 περιπτώσει τα καταφέραμε καλά, σε δύο που δεν τα καταφέραμε καταχωρήσαμε εκ νέου τις ε, πρωτοβουλίες όπως πρότεινε και το δικαστήριο. Άρα συμμορφωνόμεθα πλήρως με τις αποφάσεις του δικαστήριου. Άλλο βασικό στοιχείο που ήθελα να τονίσω είναι ότι προβλέψαμε, και αυτό αναφέρεται ήδη θετικά, προβλέψαμε λέγω για τους οργανωτές μια περίοδο τρίμηνη κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να προετοιμαστούν για να δρομολογήσουν την πρωτοβουλία. Και στην Επιτροπή προτάθηκε εξάμηνη περίοδος που ίσως να είναι κάτι παραπάνω από το αναγκαίο διότι ήδη είναι προετοιμασμένοι για την καταχώρηση. Δεν υπάρχει σαφή ζήτηση από του εμπλεκομένου φορεί από ό,τι γνωρίζουμε να παραταθεί αυτή η περίοδο στο εξάμεινο. Οπότε, εάν μετρήσετε τα πάντα, είναι 21 μήνε η όλη διάρκεια. Αν βάλουμε άλλου τρει μήνε, πάμε στα δύο χρόνια. Τι προσπαθούμε να κάνουμε για του πολίτε εκείνου που, που δίνουν ψυχή για το θέμα, να μην κρατάει περισσότερη διαδικασία από ό,τι γίνεται τώρα. Και άλλο σχόλιο για το σύστημα συλλογή στο διαδίκτυο, αν δεν το αναφέρατε ξανά. Είναι βασικό στοιχείο για μα αυτό. Θέλουμε να μειώσουμε το βάρο για του οργανωτέ, να επιτρέψουμε στου πολίτε ε, να έχουν ευκολότερη πρόσβαση και προβλέπουμε ότι αυτό πρόκειται να είναι μεγάλη βελτίωση. Και τέλο, για τι ευθύνε για την προστασία των δεδομένων. Όταν χρησιμοποιήσουμε το σύστημα αυτό στο διαδίκτυο που θα ξεκινήσει το 2020 για τη συλλογή πληροφοριών δεν θα έχουν ευθύνε για την προστασία δεδομένων και τη συλλογή στο διαδίκτυο. Σημαντικό θέμα, μειώνεται το βάρο. Και πάμε στι διάφορε τροπολογίε που υποβάλλατε για διάφορα άρθρα. Για μα, είναι η φιλοσοφία. Όλοι οι κανόνε ε, για την προστασία δεδομένων στο άρθρο 18. Διευκολύνεται έτσι το θέμα για του πολίτε και του οργανωτέ να καταλάβουν ποιε είναι οι υποχρεώσει του, ποιε είναι οι δικέ του υποχρεώσει. Αν το κατανείμουμε αυτό σε διάφορα άρθρα, ίσω να υπάρχει κάποιο κίνδυνο να επικρατεί σύγχυση για τον μέσο πολίτη, ο οποίο ε, δεν είναι συνηθισμένος ε, με νομικά κείμενα. Αυτό είναι το τελευταίο. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά ήταν η πρώτη και τελευταία παρέμβαση από αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Äh, Σας ευχαριστούμε θερμά. Ε, πέρα από το ερώτημα του τι μπορούμε να βελτιώσουμε σε οργανωτικό επίπεδο, υπάρχει και το ερώτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει λίγο παραπάνω, και το οποίο είναι τι συμβαίνει, ποια συνέχεια δίνεται σε εκείνες τις πρωτοβουλίες πολιτών που έχουν επιτυχία έκβαση. Δηλαδή, τις παραπέμπουμε κάπου, τις κάνουμε κάτι ή τελικά δεν κάνουμε κάτι. Δεν πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι όλα τα θεσμικά όργανα, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ασχοληθούμε με αυτές τις πρωτοβουλίες. Δηλαδή, θεωρώ πως οι πολίτες οι οποίοι ξεκινούν μια τέτοια πρωτοβουλία θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν το δικαίωμα αυτό του να ασχοληθούν δηλαδή τα θεσμικά όργανα με το αίτημά τους, με σοβαρότητα. Και αυτό νομίζω πως ε, ισχύει ως υποχρέωση τόσο για την Επιτροπή όσο και για το Κοινοβούλιο και για το ε, Συμβούλιο συνομοθέτες. Σίγουρα δηλαδή θα πρέπει να το έχουμε κατά νου αυτό. Γιατί αν τελικά δεν δίνεται καμία συνέχεια, δεν καταλήγει πουθενά μια πρωτοβουλία πολιτών, τελικά ε, δημιουργεί περισσότερο εκνευρισμό και περισσότερη αποξένωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί τελικά να φέρει του ε, πολίτε ε, πιο κοντά μα. Δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ απόλυτα ότι για να μειώσουμε το όριο τη ηλικία 16, εμεί προτείνουμε 5 χώρε, όχι 7. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα κάτι άλλο, γι' αυτό για του μήνες το αφήνω στην εισηγητή και το θέμα των ε, κατοίκων και της διαμονής και η απλούστευση, η εγγύηση για απλούστευση είναι τρία θέματα πολιτικά. Το πρώτο που είπαμε πριν, ε, δεν θεωρώ ότι υπάρχει καμία δέσμευση, καμία ένδειξη σαφής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δράση που θα πρέπει να δώσει μετά. Λέει ότι αυτέ που έχουν καταχωρηθεί, όλε οι συνέπειε λοιπά αναφέρονται και υπάρχουν διαπραγματεύσει και μετά θα πρέπει να προβλέπεται ένα χρόνο εντό του οποίου κάτι γίνεται. Θα θέλω να καταλάβω τον εισηγητή γιατί προβλέπει να αφαιρεθεί ένα σημαντικό σημείο του άρθρου 15. Δηλαδή, αφαίρεται η φράση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει, σύμφωνα με την άποψή του, δεν πρέπει πια να λέει ποια είναι η δράση που προτίθεται να δρομολογήσει, ή αν αλλά να λέει αν προτίθεται να παρέμβει ή όχι. Αυτό θα πρέπει να παραμείνει. Αλλιώ μειώνουμε, αποδυναμώνουμε το κείμενο και αφαιρούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υποχρέωση να πει ποια δράση θα αναλάβει, πώ θα προτίθεται να παρέμβει. Αυτή η πρόβλεψη θα πρέπει να παραμείνει κατά την απόψή μα. Ε, ευχαριστώ θερμά. Θα ξαναδώσω το λόγο στον συνάδελφο Τζαμπάσκη. Α, όχι, δεν βλέπω να θέλει το λόγο. Οπότε όλα τα υπόλοιπα θα τα διευκρινίσουμε στο πλαίσιο ε, τη συζήτηση των σχεδόν εισηγητών και στην ψηφοφορία βέβαια στη συνέχεια. 26 Μαρτίου στι 12 η ώρα είναι η προθεσμία για την υποβολή ε, των τροπολογιών και στις 20 Απριλίου θα λάβει η χώρα η ψηφοφορία. Εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία στο πλαίσιο των περιττέρων εργασιών του στον κύριο Ζαμπάτσκι και στους σκιώδεις εισηγητές. Ε, περνάμε στο τελευταίο σημείο της σημερινής διάταξης ε, της ε, δημόσιας διαβούλευσης. Εδώ πρόκειται για ε, την ε, πρόταση ε, σε ό,τι αφορά την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών. Ο κύριος Σαντιάγο είναι ο αρμόδιος συγκεκριτής μας εδώ. Η πρόθεσμη για την υποβολή των τροπολογιών είναι 26 Μαρτίου στις 4 η ώρα, ενώ εδώ στην Επιτροπή μας θα ψηφίσουμε στις 7 Ιουνίου. Αρμόδιες επί της ουσίας είναι η Επιτροπέ εμπορίου και ΙΜΚΟ. Σαντιάγο, είσαι το λόγο λοιπόν για να μα παρουσιάσει εδώ τη γνωμοδότηση. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητή Πρόεδρε. Ω ηγητή, ω συντάκτη γνωμοδότηση καλύτερα τη ε, Επιτροπή ε, Πολιτισμού και την Εισαγωγή Πολιτισμικών Αγαθών, η ΤΑΚΙΜΚΟ, είναι ε, επί τη ουσία αρμόδια. Θέλω να πω ότι ο στόχο είναι η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητε και η χρηματοδότηση της δημοκρατίας με το λαθρεμπόριο πολιτισμικών αγαθών. Και το 2008 είναι και το έτος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στόχος είναι να μην επιτρέψουμε τις αγωγές στην Ένωση πολιτιστικών μνημείων άνω των 250 ετών που παράνομα έχουν εξαχθεί από μια τρίτη χώρα. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει άδεια εισαγωγή για τι κατηγορίε αυτέ αγαθών που είναι εκτεθειμένα σε, περισσότερο, σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Θα πρέπει οι τελωνιακές αρχές του κράτους μέλους να ε, καταρτίζουν αυτή την άδεια και έπειτα για τα άλλα ε, αγαθά του παραρτήματος ε, απαιτείται η προσκόμιση απλά μιας υπεύθυνη δήλωσης από τον εισαγωγέα όπου θα λέγεται ότι έγινε νόμιμα η εξαγωγή αυτών των αγαθών από τη χώρα προέλευσής τους. Η αρχική πρόταση της Κομισιόν εισάγει μια εξαίρεση στην υποχρέωση Παροχή απόδειξη για την νόμιμη εξαγωγή από τη χώρα προέλευσή αυτών των αγαθών. Δηλαδή στην περίπτωση που η χώρα εξαγωγή, είναι δηλαδή η τελευταία χώρα που παρέμεινε το αγαθό για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να έχει υπογράψει τη σύμβαση της UNESCO το 1970, τότε απαιτείται μόνο να αποδειχθεί η νόμη από τη χώρα εξαγωγής και όχι από τη χώρα καταγωγής, από τη χώρα προέλευσης τροπολογίες μου βασίζονται στην ανάγκη να αποφύγουμε τη χρηματοδότηση παράνομων δραστηριοτήτων χωρίς να περιορίσουμε όμως με δυσανάλογο τρόπο το νόμιμο εμπόριο πολιτισμικών αγαθών. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι θα έπρεπε η υποχρέωση απόδειξης της νόμιμης εξαγωγής από τη χώρα <clears throat> προέλευσης ε, δεν είναι κάτι απαραίτητο, αρκεί να αποδειχθεί ότι ξεχθινόμε από τη χώρα εξαγωγή, γιατί συνήθω είναι δύσκολο λόγω τη αρχαιότητα και τη έλλειψη εγγράφων να αποδειχθεί σε κάποιε περιπτώσει η προέλευση του αγαθού ή σε κάποιε χώρε δεν υπάρχουν σχετικέ διατάξει που να ρυθμίζουν, να απαγορεύουν την εξαγωγή τέτοιων αγαθών. Έτσι λοιπόν να πλουστεύουμε το διοικητικό άχθο ε, και το βάρος απόδειξης. Ό,τι αφορά το, ότι το γεγονός ότι δεν εφαρμόζεται ισότιμα η σύμβαση της UNESCO 1970 από τα ε, κράτη-μέλη που την έχουν υπογράψει. Έχω να σας πω ότι δεν ε, προσφέρει λοιπόν αυτή η σύμβαση κάποια εγγύηση. Γι' αυτό όταν λέμε χώρα εξαγωγής που έχει υπογράψει, χώρα που δεν έχει υπογράψει, είναι μια διάκριση που κατά πρέπει να απαλληφθεί σε ό,τι αφορά τα 250 χρόνια αρχαιότητας για όλες τις κατηγορίες πολιτισμικών αγαθών που περιλαμβάνει το παράρτημα. Στην αρχική μου πρόταση δεν θεωρούσα ότι είναι σκόπιμο να αλλάξει, ε, αλλά το μελέτησα, το είδα ε, και σκέφτηκα μήπως θα πρέπει να ανεβάσουμε αυτό το όριο στα 500 χρόνια, γιατί <clears throat> τα αγαθά που ε, κινδυνεύουν να, να κλαπούν να, ή να υποστούν βεβήλωση οτιδήποτε άλλο είναι πράγματι τα πιο πολλά πάνω από 500 ε, χρόνια ε, πάνω από 500 ετών βέβαια θα πρέπει γενικά να προστατεύσουμε τα πληθυντικά αγαθά τρίτον επειδή το κείμενο της Κομισιόν προβλέπει εξαίρεση στο παιδί εφαρμογής της οδηγίας όταν είναι εκπαιδευτική, επιστημονική ή σκοπή ή ακαδημαϊκής έρευνας, θα έπρεπε πιστεύω εδώ να συμπεριλάβουμε και τα έργα αποκατάστασης, ανάπλασης. Το αρχικό κύμα της Κομισιόν επίσης θεωρεί το να μπορεί ένα αγαθό να εξάγεται μόνιμα, μάλλον θεωρεί την περίοδο του ενός μήνα ως permanent μόνιμο. Αν δεχθούμε την πρόταση όμως, να μην ε, αποδεικνύεται η νόμιμη εξαγωγή από τη χώρα προέλευσης, θα έλεγα για να έχουμε νομική ασφάλεια, να καταργήσουμε και αυτή την διάταξη περί ελάχιστης ε, παραμονής του αγαθού. Τώρα, οι τελωνιακές αρχές, εφόσον το θεωρούν σκόπιμο, θα μπορούσαν να απαιτούν πρόσθετες πληροφορίες και να εξετάζουν τα ίδια τα αγαθά. επειδή είναι μια ιδιαίτερη ε, μορφής αυτά τα αγαθά, νομίζω ότι αυτό που είναι απαραίτητο είναι να, αγγίσουμε, να αγγιθούμε την αποθήκευσή τους σε κατάλληλες αποθήκες, σε κατάλληλους χώρους. Επίσης, για να ε, διευκολύνουμε την πρόσβαση στα νέα συστήματα και για την ε, εκπαίδευση και κατάρτιση των αρχών και των επαγγελματιών που οργανώνουν τα κράτη-μέλη και για να προωθήσουμε και εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τους αγοραστές προτείνω να υπάρχουν σημεία επαφής και ενημέρωση κάθε κράτος μέλος. Τέλος, πρέπει να ενισχυθεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση με ηλεκτρονικά έγγραφα, ε, τυποποιημένα έγγραφα για της άδειε εξαγωγής, αγωγής ή τα έγγραφα <clears throat> της βεβαίως πρέπει να, παρέχουν, ε, να παρέχονται στις ελληνικές αρχές ώστε να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος επίσης του forum shopping. Θα πρέπει να είναι ομοιόμορφες αυτές τις διαδικασίες. Δεν θα πρέπει επίσης να μας διαφεύγει ποιος είναι ο βασικός στόχος. Είναι η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης του λαθρεμπορίου ε, τέτοιων πολιτικών αγαθών ε, για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και όχι η προστασία των πολιτικών αγαθών εν Αυτά είχα να πω. Περιμένω να συνεργαστώ πολύ καλά με τους συναδέλφους για να πετύχουμε το διπλό στόχο, κατά πολέμηση της παράνομης, μάλλον, για να καταπολεμήσουμε τρομοκράτηση της τρομοκρατίας και να εξασφαλίσουμε και την αποτελεσματική προστασία τη πολιτισμική κληρονομιά. Yeah, σε ευχαριστούμε Σαντιάγο. Λουίτζι Μόργανο. Ευχαριστώ. Από την πολιτική μου ομάδα πρέπει να πω ότι συμφωνούμε όσον αφορά τον επιδιωκόμενο στόχο του εισηγητού. Μετά πρέπει να εξετάσουμε την ουσία των θεμάτων. Θα είχα πολλά να πω, διότι θεωρώ ότι η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη από ό,τι περιεγράφει. Θα συνοψίσω βασικά σημεία και μετά θα προτείνω και τροπολογίες σχετικές. Όπως είπε ο εισηγητής, είναι κατεπίγουση ανάγκη θέσπιση αποτελεσματικών μέτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιταχθούμε στις παράνομες αγωγές πολιτιστικών αγαθών, μεταξύ των οποίων το λαθρεμπόριο αντικειμένων αρχαιοτήτων που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και όχι μόνο γι' αυτό χρειάζονται συγκεκριμένα οι φορείς για κάτι τέτοιο. Έχουμε, πρέπει να έχουμε ιδιαίτερα σώματα που θα ασχολούνται με το θέμα αυτό, κρατικούς φορείς. Και θα πρέπει να προβλέπεται και αποκλεισμό των εισαγωγών ή το εμπόριο όταν προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές αυτά τα αγαθά. Διαφορετικά άλλα θα λέμε και μετά δημιουργούνται εμπορικά τρίγωνα. Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνει αυτό εμείς είμαστε η Επιτροπή Πολιτισμού και πρέπει να γραμμίσουμε και κάτι που μας ανήκει σαν πτυχή. Αλλιώς γιατί σχολούμεθα. Πρώτη πτυχή. Δεν πρέπει να ζημιώσουμε μέσω διαφόρων επιχειρήσεων άμεσα την ιστορική, πολιτισμική και αρχαιολογική κληρονομιά των χωρών προέλευσης. Και πολύ συχνά το συζητούμε αυτό. Το πρόβλημα είναι να κάνουμε το καθήκον μας. Το 2018 είναι Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Δεν είναι μόνο δικό μας, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και σε αυτή την κατεύθυνση. Να το πω ειλικρινά, όσον αφορά την πρόταση, έχουμε διάφορα σημεία επίκριση. Και όσον αφορά αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη, όσον αφορά την πρόταση του συγητού. Όσον αφορά την πρώτη πτυχή, συμφωνώ με τον εισηγητή, με την πρόταση που κάνει. Να έχουμε πληροφορική που θα χρησιμοποιούμε για τη διαδικασία, να μπορούν να χρησιμοποιούν διαδικτυακά μέσα και θα μπορούν τελωνιακές αρχές να ανταλλάσσουν ε, ταχαίως τις πληροφορίες. Οι υπηρεσίε πολιτισμού και των τελωνίων ανταλλάσσουν πληροφορίε γρήγορα στα κράτη-μέλη. Χρειάζονται εκστρατείε ευαισθητοποίηση, κυρίω όσον αφορά του αγοραστέ να ενημερώνονται. Και μετά χρειάζονται και θηρίδε πληροφόρηση ενημέρωσης. Επανειλημμένα αναφέρθηκε μια ιδέα από τον εισηγητή. Είπε να ξεπεράσουμε την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ...το άρθρο 4, να διαφοροποιήσουμε την περίπτωση όπου η εξαγωγική χώρα έχει υπογράψει τη σύμβαση της UNESCO. Αυτό το καταλαβαίνω. Αν το αφαιρέσουμε αυτό, Πώς καθορίζουμε τη χώρα προέλευσης. Εξαλείφουμε τον ορισμό της χώρας προέλευσης. Γιατί το λέω αυτό. Έχουμε 134 χώρες σήμερα που έχουν υπογράψει τη συνθήκη της UNESCO, τη σύμβαση της UNESCO. Για ποιες χώρες δεν θα κάνουμε κάτι τέτοιο. Ε, τι φόβος κρύβεται πίσω από αυτή την πρόταση. Τι δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε σαν θέμα. Κατά την άποψή μου, εμείς θα πρέπει να επιλέξουμε την αντίθετη προσέγγιση διότι βασική αναφορά της νομοθεσίας πρέπει να είναι η χώρα προέλευσης, σύμφωνα με τη σύμβαση της UNESCO. Το να μην αναφέρουμε τη σύμβαση της UNESCO σημαίνει ότι δεν θέλουμε να προστατεύσουμε αυτό το στοιχείο. Και νομίζω ότι αυτό είναι αντιφατικό. Θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στο πολιτιστικό αγαθό, άρθρο 2. Αυτό μας αφορά σαν Επιτροπή. Έχουμε αρμοδιότητα μαζί με την ΙΤΑ και ΙΝΚΟ πάνω σε αυτό. Δώστε μου άλλα δύο λεπτά παρακαλώ. Γιατί το λέω αυτό. Όσον αφορά τον ορισμό, υπάρχει το ελάχιστο όριο 250 έτη για το αγαθό. Λέω εισηγητή θέλει να το πάει στα 500. Εγώ πρέπει να πω ότι που δεν συμφωνούμε. Το όριο 250 και όχι των 500 που δεν υπάρχει πουθενά δεν έχει χρησιμοποιηθεί για καθορισμό πολιτιστικού αγαθού. Αυτά τα 250 χρόνια δεν σέβεται καμία διεθνή συνθήκη. Και το αναφέρω γιατί θα υποβάλουμε σχετικές τροπολογίες. Τη Σύμβαση της Χάγης για την προστασία της πολιτιστικής ιδιοκτησίας σε περίπτωση ένοπλης σύραξη. Φερρυπίν. Άρθρο 1. Σύμβαση για τα μέσα παγόρευσης εισαγωγής παράνομης μεταφοράς εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών. Το 70. Σύμβαση για τα πολιτιστικά αντικείμενα που κλέπτονται και εξάγονται παράνομα. Άρθρο 2. Επίπεδο διεθνών συμβάσεων. Ε, έχουμε 50, 70 και 100 έτη. Στην UNESCO δίνουμε 70. Και λέω ότι το πεδίο εφαρμογή είναι κάτω από τα 100 έτη. Αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να συνεννοηθούμε. Γιατί, αν πάμε στα 250 χρόνια, πάμε κινηματογράφος, μουσική, γραμματόσημα, καταγεγραμμένη μουσική. Ε, τι γίνεται. Και είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα αγαθά. Έχουμε πολιτικό στόχο να θέσουμε. Την προτεραιότητα της Επιτροπής Πολιτισμού. Πολιτική προτεραιότητα να εγγυηθούμε. Διακόπτη, Πρόεδρος. Λουίτζι, ήμουν γενναιόδορη, αλλά τελικά έχει πάρει το λόγο για περισσότερο από ότι ο ίδιο ο εισηγητή. Δεν μπορώ να το επιτρέψω, συγγνώμη. Έλγα Τρούπελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πέτρα, και ευχαριστώ τον Σαντιάγο για αυτή την παρουσίαση τη ε, έκθεση. Ε, δεν είναι η πρώτη φορά που συζητούμε αυτό το δύσκολο ζήτημα εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού. Και όταν λέω δύσκολο, εννοώ από την άποψη τη επίλυσή του. Δηλαδή, λαμβάνουμε υπόψη μα όλα τα ζητήματα, τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία, τη χρηματοδότηση κάποιων πολύ ανητικών συμπεριφορών σε χώρες όπου από τη μία πλευρά καταστρέφουν πολιτισμικά μνημεία, ενώ από την άλλη πλευρά προσπαθούν να εξαγάγουν τέτοια πολιτιστική κληρονομιά. Δηλαδή σε χώρες όπου δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για την ε, πολιτιστική ε, ε, και ποικιλομορφία αλλά και την συντήρηση ε, του πολιτισμού και ό,τι καθεξής. Άρα λοιπόν εμείς από την πλευρά της Ευρώπης θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί κάτι τέτοιο άπτεται των βασικών μας τον και του κράτους δικαίου και των βασικών μας αξιών. Άρα λοιπόν είναι πολιτική μας ευθύνη να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάχρηση των αγορών έργων τέχνης. Γιατί αν δεν είμαστε, αν δεν επαγρυπνήσουμε, τότε θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ θα καταστούμε μέρο, αν θέλετε, αυτής της, αυτού του συστήματο κατάχρηση των έργων τέχνης. Ε, απλώς και μόνο για, ε, για κερδοσκοπία. Αναφερθήκαμε σε αυτό το ζήτημα της σύμβασης της UNESCO και της ε, χώρες ε, προέλευσης. Ε, νομίζω πως αυτό που αναφέρεται από τον Σαντιάγο είναι σημαντικό. Δηλαδή ακόμα και εν ώψη και των ε, ευρωεκλογών είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό να προλάβουμε να έχουμε έναν κανονισμό σε ό,τι αφορά τα έργα τέχνης και την εμπορία τους. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Σίλβια. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο Φίσα. Εντάχει. Διότι πολλά είπε και ο συνάδελφος Μόργανο. Εκφράσω ανησυχίες στην πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά την άποψή μου, υπάρχει μια αλληλεπικάλυψη μεταξύ ενός θέματος πριν της εναρμονίσεως των κανόνων εισαγωγής εν γέννη και του θέματος του ειδικού ενδεχόμενου λαθρεμπορίου και χωρών σε σύραξη. Όλα πάνε μαζί. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Τα 250 χρόνια. Σύμφωνα με αυτό που είπε ο κ. σε καμία διεθνή σύμβαση δεν υφίσταται περίοδος άνω των 100 ετών. Κάτω των 100 ετών μάλλον. Νομίζω ότι από την πλευρά του κανονισμού λείπει αναφορά στους δύο φυστάμενους κανονισμούς. Μετά την σύγκρουση Συρία και στο Ιράκ. Στις χώρες αυτές δεν αναφέρονται οι χώρες σε σύραξη. Αυτές που είναι σε σύραξη. Ήδη αποφάσισε το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον αποκλεισμό εισαγωγών ε, από χώρε που είναι σε σύραξη. Ή βοήθεια, δίνεται βοήθεια ε, να, να επανακτήσουν τα αγαθά τους ή να τα αποκαταστήσουν τα πολιτιστικά αγαθά. Και δεν υπάρχει αυτό. ενώ στην πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορούμε να το καλύψουμε ίσως. Άλλο σημαντικό. Δεν μιλάμε ποτέ για το θέμα της κατάρτισης. Τη στενή διασύνδεση μεταξύ τελωνιακών αρχών και πολιτιστικών αρχών, κάτι που υπάρχει στη χώρα μας. Πρέπει να αναφέρεται. Αναφέρουμε και κάτι άλλο. Θα πρέπει στα κάτι μελη να θεσπίσουν μονάδες ειδικέ για καλύτερη εξυχνίαση υποθέσεων, ανταλλαγή πληροφοριών και κοινή παρέμβαση. Ελάχιστα αναφέρονται πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά. Η Ζαμίνα Φαχάν έχει το λόγο. Ευχαριστώ θερμά τον Σαντιάγο για αυτήν την πρόταση εκθέσεως η οποία βέβαια θα τροποποιηθεί με βάση τροπολογίες που θα υποβληθούν. νομίζω πως αυτό που κατέστη ε, σαφές από όλες τις παρεμβάσεις είναι ότι ο βασικός μας στόχος θα πρέπει να είναι η καταπολέμηση, η πρόληψη της εισαγωγής πολιτισμικών αγαθών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εντάξει, αναφέρθηκε ενίοτε το ζήτημα της εξαγωγής τέτοιων αγαθών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα δεν είναι εξαγωγή. Έχουμε πολύ σαφείς κανόνες σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές τέτοιων αγαθών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα είναι η εισαγωγή τους. Εάν θέλουμε λοιπόν ή αν τελικά το αποτέλεσμα είναι να περιπλέξουμε ακόμα περισσότερο το κανονιστικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά την εμπορία των πολιτιστικών αγαθών, δεν μπορεί να είναι κάτι τέτοιο προ όφελο μα. Δεν θα πρέπει δηλαδή τελικά να καταστήσουμε από ρεαλιστική άποψη αδύνατη μια αποτελεσματική εμπορία ε, πολιτισμικών αγαθών. Αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε είναι παράνομη εξαγωγή τέτοιων αγαθών και στη συνέχεια εισαγωγή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αυτό που θα πρέπει να καταπολεμήσουμε είναι ότι δεν θα εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αγαθά πολιτισμικά τα οποία προέρχονται από, ε, που έχουν εξαχθεί παράνομα από άλλε χώρε, για παράδειγμα που βρίσκονται σε πόλεμη ε, σύραξη. σε περιπτώσεις δηλαδή όπου υπήρξε κλοπή, αρχαιοκαπηλεία ή έχουν αφαιρεθεί από ένα συγκεκριμένο σημείο ορισμένα αγαθά χωρίς ε, να επιτρέπεται κάτι τέτοιο, σίγουρα θα πρέπει να μην είναι δυνατόν να έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε ό,τι αφορά την ε, αρχή της χώρας προέλευσης δεν ισχύει πάντοτε, γιατί θα πρέπει να δούμε τελικά, εάν για παράδειγμα βρίσκεται ένα πολιτισμικό αγαθό σε μια χώρα προέλευση, το οποίο όμω έχει για παράδειγμα εξαχθεί παράνομα από άλλη χώρα καταγωγή εκεί. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα παρακολουθειται η εμπορία ενός πολιτισμικού αγαθού. Ε, πάντως, επί της αρχής, νομίζω πως ε, αυτό που προτείνει ο Σαντιάγο, δηλαδή αρχή της χωρα ε, χώρας εξαγωγής, επαρχεί ε, για τους σκοπούς μας. Ευχαριστώ, λέει πρώτος. Δεν ξέρω αν ο εκπρόσωπος της Επιτροπής θέλει να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σύντομα, δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα, καλωσορίζουμε το γεγονός ότι φαίνεται θετικά να ε, αντιμετωπίζετε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δύο σημεία κυρίως μας προκαλούν κάποια ανησυχία. Το πρώτο είναι η όλη συζήτηση για τα 250 ή 500 έτη minimum. Νομίζω ότι στην πρότασή μας προσπαθούμε να υπάρξει μια ισορροπία που να σέβεται την ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς αφενός, αλλά και την αποφυγή υπερφόρτωσης των ε, αρχών με διοικητικό βάρος αφετέρου. Άρα 250 minimum νομίζω ότι είναι μια ενδεδειγμένη λύση και βασίζεται ε, σε λύσεις που φαίνεται να αποδίδουν άλλους στον κόσμο. Επίσης, σε ό,τι αφορά ένα άλλο θέμα. Source ή export country. Δηλαδή χώρα προέλευσης ή χώρα εξαγωγής. Αυτό που ενδιαφερόμαστε εδώ είναι να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της χώρας προέλευσης. Source country. Και θα πρέπει να λαμβάνονται αυτά τα συμφέροντα υπόψη στη λύση που θα βρούμε και να μην δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου θα μπορούν εύκολα οι κανόνες να παρακάμπτονται. Άρα να είναι καινογράμμα οι διατάξει αυτέ. Σημείωσα ε, πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες και από πλευρά μα είμαστε διατεθειμένοι να συνεισφέρουμε εμεί στην περαιτέρω και πολιτική και τεχνική συζήτηση που θα διεξαχθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Σαντιάγο, άλλη μια φορά τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα με πολύ προσοχή τις προτάσεις των συναδέλφων. Φυσικά, όταν μίλαγα για 500 χρόνια εγώ, το έλεγα πώς να το πω, ως ιδέα προς μελέτη, προς εξέταση, δεν ήταν πια και γραμμένο σε μάρμαρο, μπορεί να είναι 150, μπορεί να είναι 100, μπορεί να είναι 500. Αυτό προσπαθούμε εμείς να κάνουμε εδώ είναι να ρυθμίσουμε όχι την εισαγωγή οποιοδήποτε πολιστικού αγαθού. Απλά δεν θέλουμε τα αγαθά αυτά να χρησιμοποιηθούν ε, για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως είπα. Φυσικά με ένα γραμματόσημο δεν θα χρηματοδοτηθεί η τρομοκρατία, αλλά με τη διακίνηση ε, αρχαιοτήτων σε που, από χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο. Και αυτά τα, ε, αυτές οι αρχαιότητες σίγουρα είναι πάνω από 500 ετών. Εγώ απερίφραστα επιμένω στο ότι πρέπει να έχουμε μια προθεσμία. Τώρα το αν θα είναι 500 χρόνια, ή αν θα είναι 400, θα το δούμε. Τώρα σε ό,τι αφορά ε, τις εισαγωγές από χώρε που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Ε, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το μελετήσουμε ακριβώς πώς θα διατυπώσουμε τη σχετική διάταξη. Το είπε και η Σαμπίνε. Το θέμα είναι να μην περιπλέξουμε την νόμιμη εισαγωγή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ μίλησα με πολλούς ε, αντικέρ ε, και με ενώσεις, όπως πέραν χάρη ε, από τη Γερμανία μια ένωση για τα παλαιά νομίσματα. Και μου είπαν ότι ναι, πρέπει να προσπαθήσουμε να συμφιλιώσουμε όλα αυτά τα θέματα. Αυτό που πρέπει όμως να είναι προτεραιότητα είναι πώς θα καταπολεμήσουμε το λαθρεμπόριο πολιτικών αγαθών που χρησιμοποιείται μετά για χρηματοδότηση τη δημοκρατία, αλλά και πώς δεν θα παρακολύσουμε ταυτόχρονα το νόμιμο εμπόριο πολιτικών αγαθών. Και έχουμε και το θέμα του κόστου ε, των εισαγωγών που δεν θα πρέπει να αυξηθεί δυσανάλογα. Επίση, πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ ταλωνιακών αρχών και πολιτιστικών αρχών των διαφορών χωρών. Θα πρέπει επίση να υπάρξει εκπαίδευση των εμπειρογνωμόνων, των ειδικών τελωνιακών υπαλλήλων και ευαισθητοποίηση βέβαια και τη κοινή γνώμη για το θέμα αυτό. Είμαι στη διάθεση των συναδέλφων να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και είμαι αισιόδοξο ότι θα καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική λύση που θα πρέπει να μα δώσει τη δυνατότητα να αποφύγουμε το λαθρεμπόριο και τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία πάνω απ' όλα, αλλά ταυτόχρονα να μην επιβάλλουμε υπερβολικά προσκόμματα στο νόμιμο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών. vielen herzlichen Dank. Ich glaube, die Diskussion... Σας ευχαριστώ θερμά. Νομίζω πως η συζήτηση κατέδειξε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό φάκελο όπου ε, το ζητούμενο είναι να διατηρήσουμε και την κατάλληλη ισορροπία. Δηλαδή από τη μία πλευρά να αποτρέπουμε παράνομες εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς από την άλλη πλευρά να καταστήσουμε αδύνατο ε, το εμπόριο με αυτά τα αγαθά ή χωρίς τέλος να το επιβαρύνουμε με υπερβολικές ε, γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ε, πεπισμένο ότι οι σχέδιοι ε, και οι σχέδιοι θα, ε, θα φτάσουν σε ένα καλό αποτέλεσμα. Όπως είπαμε, 26 Μαΐου στις 4 το απόγευμα η προθεσμία για την υποβολή συνόμη των τροπολογιών και 7 Ιουνίου η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Τώρα φτάσαμε στο τέλος της δημόσια διαβούλευση. Έχουμε ένα ακόμα σημείο στην ημερήσια διάταξη και κλεισμένο των θυρών. Οπότε όσοι δεν είναι μέλη του Κοινοβουλίου εδώ θα ήθελαν να εγκαταλείψουν την αίθουσα έτσι ώστε να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μα και κλεισμένο όπω είπα των θυρών. Και επίση ζητώ να σταματήσει το web streaming τη συνεδρίαση.